μετά από την διακοπή τη συνεδρίαση χθε το βράδυ, επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διαταξή μα είναι η παρουσίαση από το Συμβούλιο του Σχεδίου του Γενικού Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2010. Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τον κύριο Hans Lindblad από την πλευρά του Συμβουλίου. Είναι ο Υφυπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Σουηδίας. Χαιρετίζω επίσης την παρουσία του κυρίου Αλγκέρντας Σέμετα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω και τα δύο σώματα για την παρουσία τους στη σημερινή συνεδρίαση και δίνω μέσα στο λόγο στον κύριο Λίντεπλατ, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά είμαι ενώπιόν σας και είναι μια μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας παρουσιάσω το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Καταρχήν την οικονομική κατάσταση η οποία επικρατεί, η οποία έχει ανησυχητικό χαρακτήρα Πολύ περισσότερο βέβαια πριν από έξι μήνες από ότι σήμερα που τα πράγματα φαίνεται να σταθεροποιούνται. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχουν μειωθεί. Αντιμετωπίζουμε όμως παρόλα αυτά προβλήματα όπως είναι η ανεργία, τα προβλήματα στις χρηματαγορές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προβλέψουμε μακροπρόθεσμα για τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης με έναν τρόπο που θα είναι σταθερός και αηφόρο. Πολλές χώρες έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διατρέξουν για να επιτύχουν τη χρηματοοικονομική ισορροπία. Επίσης η δημογραφική εξέλιξη θα έχει επιπτώσεις για τα δημοσιονομικά μας όπως και οι κλιματολογικές αλλαγές οι οποίες μας υποχρεώνουν να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να κατανέμουμε τα δημόσια κονδύλια. Επίσης, είναι απαραίτητο να δείξουμε σοφροσύνη και προσοχή για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προσθέμενη αξία την οποία μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο την ε, κρίση στιγματοοικονομική και συγγνώμη έπρεπε να είχα σηκωθεί για να μιλήσω δεν είμαι πολύ ψηλό, αλλά φαίνεται πρέπει να σκύβω για να μιλάω στο μικρόφωνο Πρέπει να ενισχύσουμε επίση την μακροπρόθεσμή μα ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεται μια ενιαία δράση από όλου μα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει με ένα προπολογισμό ο οποίο υπόκειται σε πειθαρχία και να αντιμετωπίσουμε θέματα όπω είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, να δημιουργήσουμε υποδομέ, να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα και να ενθαρρύνουμε την συνοχή στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προσπαθεί να πράξει το Συμβούλιο μέσα του σχεδίου προπολογισμού. Η λογική που διέπει το σχέδιο προπολογισμού είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ε, απασχόληση, την ευμάρεια στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εδραιώσουμε μια πολιτική η οποία θα είναι αξιόπιστη, μια πολιτική η οποία θα είναι σταθερή και αηφόρο και εφικτή φυσικά, δίνοντα την έμφαση στι απαραίτητε ε, υποδομέ ώστε να είναι σταθερή αυτή η οικονομία και να εξασφαλίσουμε και την ισότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχο λοιπόν του σχεδίου μα είναι να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία, αλλά επίση να είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση με τον προπολογισμό του 2009. Αυξάνουμε τι πιστώσει πληρωμών όπω και τι πιστώσει υποχρεώσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η πρότασή μας ως μια αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον και την επίτευξη ορισμένων στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα μια ταχεία απάντηση στι προκλήσει αυτέ. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα εκεί που η Ευρώπη μπορεί να δώσει μια, μια προσθέμενη αξία. Η λιτότητα του προπολογισμού και η σταθερότητα τη διαχείριση είναι απαραίτητε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον ισολογισμό των δημοσίων οικονομικών τη Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό επίση να σεβαστούμε τι οροφέ των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι απαραίτητο όμω επίση να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη ε, ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε καταστάσει οι οποίε καταρχήν μπορεί να είναι απρόβλεπτε. Το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει 108 ε, εκατομμύρια 38 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών και περιέχει μία σειρά από δράσεις οι οποίες έχουν λάβει υπόψη την δυνατότητα εφαρμογής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ικανότητα απορρόφησης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την ανάλυση του Συμβουλίου. Θέλω τώρα να κάνω μια επισκόπηση των κεφαλαίων. Στο τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, εδώ δίνουμε έμφαση στην ενέργεια, στις ε, ενεργειακές υποδομές. Και όλα αυτά Μα δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό στο τομέα αυτό κατά 8%. 8% είναι ένα σημαντικό ποσό. Όπως γνωρίζετε, όλα αυτά θα χρηματοδοτηθούν και μέσω του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης και αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν μέσα στο φθινόπωρο. Για το κεφάλαιο 1β, το Συμβούλιο ενστερνίζεται τις προτάσεις της Κομισιόν για τον τομέα των πληρωμών θεωρούμε ότι μπορούμε να επιφέρουμε κάποιε περικοπέ σε σχέση με την αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το σχέδιο προπολογισμού, μα σημαίνει και μια αύξηση τη πιστώση πληρωμών κατά 3,2 σε σχέση με το 2009. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 2, εκεί το Συμβούλιο προτείνει μια σημαντική αύξηση τόσο σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, όσο και για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. 4,9% για τις πιστώσεις ε, δέσμευσης υποχρεώσεων. Και στο κεφάλαιο 3 έχουμε κάποιες μικρές ε, διαρρυθμίσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν εδώ. Θα υπάρχουν επαρκείς ε, πόροι για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μετανάστευσης και την Frontex για το κεφάλαιο 4. <clears throat> Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε ένα επαρκές περιθώριο στο κεφάλαιο αυτό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν όλος απρόοπτος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προβλέπουμε ένα περιθώριο περίπου 310 εκατομμύριων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Αυτό για μας είναι κεφαλαιόδες αν θέλουμε πραγματικά να καλύψουμε τα απρόβλεπτα αυτά. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό για την ε, κατεπίγουσα βοήθεια και αρρωγή, εκεί δεχόμαστε ακριβώ την πρόταση τη Κομισιόν. Επίση, για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, τα ποσά τα οποία προβλέπονται φέτο έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι για να έχουμε την απαραίτητη ικανότητα. Κεφάλαιο 5. Τώρα διοικητικέ δαπάνε. Εδώ είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με τρόπο πλήρη, ο στόχος μας είναι οι διοικητικέ δαπάνες να μην αυξάνουν ταχύτερα από τον ρυθμό πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αντανακλάται και στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπουμε λοιπόν οι δαπάνες οι διοικητικέ να παραμείνουν περίπου σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο και σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη την διεύρυνση του 2004 και του 2007, να λάβουμε υπόψη την ανάγκη πλήρους τελέχωσης στις νέες θέσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί στα οργανογράμματα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προηγούμενη Προεδρία το είχε τονίσει εξάλλου ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα γίνει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο η πρόσληψη νέων υπαλλήλων για όλου του υπαλλήλου και είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό και θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου για τα θέματα αυτά. Πρωτού κλείσω. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας τον Ιούλιο ήταν πολύ καλή το κλίμα το οποίο επεκράτησε και νομίζω ότι μόνο με ένα τέτοιο καλό κλίμα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Συνήθως είναι πολύ σύντομες ομιλίες του Συμβουλίου και οπότε μας εκπλήξατε και ε, παρακαλώ και εγώ πειθαρχώ σε αυτού του κανόνε. Επομένω, θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε αυτά τα χρονικόρια τα συνήθεια τα οποία υπάρχουν. Οπότε, ε, αυτά και σα ευχαριστώ και πάλι για την εισήγησή σα. Στα πολωνικά τώρα, ε, ο επόμενο. Θα είναι ο κύριο ε, Σέμετα εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά μου δίνετε αυτή η ευκαιρία σήμερα το πρωί να απευθύνω τον λόγο σε όλου εσά και γνωρίζω ότι οι πρώτε φάσει τη διαδικασία του προπολογισμού, ιδίω όσον αφορά την συνδιαλέγη τον Ιούλιο, έγιναν υπό ε, μια συγκυρία μάλλον θετική και ελπίζω ότι θα έχει την ίδια συνέχεια ε, η συνεργασία μα για τι αμέσω επόμενε εβδομάδε. Ακόμα έχουμε δουλειά μπροστά μα μέχρι να ολοκληρώσουμε τον προπολογισμό και έχουμε ακόμα κάποια ζηματικά θέματα τα οποία κρεμούν, όπω η δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν ε, με τρόπο επικοδομητικό. Μετά την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο, αφού αποφασίστηκε το σχέδιο προπλησμού του χρήση του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι οι προτάσεις του Συμβουλίου είναι θετικότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις που θα πρέπει να σας αναλύσω. Δυστυχώς 1,8 δις ευρώ ε, περικόψαν από το Συμβούλιο όσον αφορά τις πιστώσεις των πληρωμών. Και αυτό έχει σημασία για το 1α και για το κεφάλαιο 4. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό όσον αφορά την απασχόληση, όσον αφορά την ανάπτυξη και όσον αφορά επίσης την αρρωγή ε, στην προενταξιακή φάση προς άλλες χώρες. Επίσης, έρευνα, διοικητικά, διοικητικές δαπάνες και εκεί είχαμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές περικοπές. Θα πρέπει μας να ληφθεί υπόψη το τι ισχύει για κάθε περιφερειακή υπηρεσία. Ε, άρα να γίνεται κατά περίπτωση η αντιμετώπιση κάθε περιφερειακής υπηρεσίας και μην έχουμε οριζόντιες περικοπές για όλους. Επίσης, στην έρευνα και στις εξωτερικές ε, δράσεις και εκεί θα πρέπει να δούμε τα προγράμματα πώς θα πρικοδοτηθούν όπως πρέπει. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα φροντίσει τόσο ώστε να, ε, να αντισταθμιστούν αυτές οι περικοπές του Συμβουλίου, ιδίω για το 1α και για το 1β, όσον αφορά επίσης τις πιστώσεις πληρωμών και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει το Συμβούλιο ότι υπάρχουν ευξημένες ανάγκες στην Γεωργία ε, και εμεί θα υποβάλουμε σχετικέ μα προτάσει τέλο Οκτωβρίου. Μέχρι σήμερα έχουμε υποβάλει στην αρχή επί του προπολογισμού μια διορθωτική επιστολή ώστε να ε, επικαιροποιήσουμε το κεφάλαιο 4. Εδώ χρειάζονται 95, ευρώ, 95 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω και άλλα 60 ευρώ παραπάνω ε, σε πληρωμές και υποχρεώσεις αντιστοίχως όσον αφορά την Παλαιστινιακή Αρχή και όσον αφορά την ενοικοδόμηση της Λωρίδας της γάζης. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι συνοδευτικά μέτρα θα γίνουν ούτως ώστε να δούμε τι εμπορικές συμφωνίες θα συναυθούν για να δούμε ε, πώς θα βοηθήσουμε τις ε, μπανανοπαραγωγές χώρες της ΑΚΕ. Επίσης 50 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να διατεθούν όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικουρήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μία ε, αγαστή συνέχεια, ε, μια επιτυχημένη συνέχεια στη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Σε σχέση με τον τίτλο ή κεφάλαιο 5, εμείς δεν ζητήσαμε πάρα πολλά στο προσχέδιο του προπολογισμού ή στο σχέδιο του προπολογισμού και είπαμε ότι θέλουμε μόνο 0,9% ε, αύξηση σχέση με τη χρήση του 2009 όσον αφορά τις διοικητικές δαπανές τις δικές μας. Ε, όμως, το Συμβούλιο δυστυχώς περιέκοψε ακόμα περισσότερο τις ε, δικές μας ε, διοικητικές ε, δαπάνες για την επόμενη χρήση. Εν κατακλείδη, ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκαταστήσει την τάξη όσον αφορά αυτέ τι περικοπέ και ελπίζουμε ότι θα είναι επικοδομητικέ οι συνομιλίε μεταξύ των τριών οργάνων και τελικά θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια αίσια κατάληξη όσον αφορά την διαδικασία, την δημοσιονομική και την φετινή. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σέμετα όσον αφορά τι δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Επίσης, ευχαριστούμε γιατί και εσεί εσείς στηρίσατε το χρονικό όριο για την αγόρευση το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων που είναι στην αρχή τη φάση, διότι η κυρία συζήτηση θα γίνει σε λίγε εβδομάδε αφού λάβουν χώρα οι ε, ζυμώσει στην Επιτροπή των Προπολογισμών. Και τώρα αρχίζουμε από του ε, αρμόδιου ε, εισηγητέ. Πρώτο ο κύριο Λάβλο Σούριον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, θα μιλήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα, στα Ουγγρικά. Και αυτό είναι ένα αυτονόητο δικαίωμα να χρησιμοποιεί κανείς τη μητρική του γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα επίσημα όργανα της. Κανείς δεν μπορεί να περιορίσει αυτό το δικαίωμα. Εγώ ήλπισα ότι η οικονομική κρίση θα οδηγούσε σε μια αντιμετώπιση για να υπάρξει ανάκαμψη και αύξηση της απασχόλησης, αλλά συγχρόνως ότι θα παρήχε και μια θετική ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθμισε τη θέση του τον προηγούμενο Φεβρουάριο και την συνέδεσε τη θέση του με τις ελπίδες ότι το, το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν θα ακολουθούσαν την ίδια γραμμή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά βλέπουμε ότι μεγάλα μέρη αυτής της πρότασής μας δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση του προϋπολογισμού. Το τμήμα εσόδων του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι ένα μεγάλο άχθος για τα κράτη-μέλη και ούτω ή άλλω τα κονδύλια αυτά δεν είναι επαρκή για την επίτευξη των στόχων. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του προπολογισμού που πηγαίνει στη Γεωργία, παρόλα αυτά οι Γεωργοί μας διέρχονται μια πολύ μεγάλη κρίση ένα μεγάλο μέρος της ε, χρηματοδότηση του προπολογισμού είναι η πολιτική συνοχή. Παρ' όλα αυτά αυξάνονται συνέχεια οι ανισότητε μεταξύ των περιοχών τη Ευρώπη, αντί να μειώνονται. Ελπίσαμε στο παρελθόν ότι η κρίση αυτή θα ήταν μια ευκαιρία να αυξήσουμε τα κονδύλια στον τομέα τη έρευνα και τη κοινοτομία και στην καλύτερη ε, κατανομή των κονδυλίων του προπολογισμού ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό ο προπολογισμό αυτό. Επίση είχαμε ελπίσει ότι ο προπολογισμό αυτό. θα χρησιμοποιείται με ένα τρόπο ο οποίος θα είναι ορθός και χριστός, χωρίς διαφθορά σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων, αλλά ελπίσαμε επίση ότι και τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και προσθέμενη αξία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στοχεύσει ο προπολογισμό αυτό να αποτελεί ένα σαφέ μήνυμα προ του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα που προέρχονται από την οικονομική κρίση και να αυξηθεί η προσθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε φυσικά και τι δικέ μα προτάσει για το πώ θα αναζωογονήσουμε και πάλι την οικονομία τη Ευρώπη. Επίση, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Και εδώ η ελπίδα μα ήταν όχι μόνο να υπάρχουν μερικά ειδικά προγράμματα τα οποία καλύπτονται από λίγα εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση τη κρίση, αλλά ελπίζαμε ότι σε όλε τι γραμμέ του προπολογισμού θα ακολουθείται ο στόχο τη αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο προπολογισμό στην υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τώρα ο κύριος Βλάντιμιρ Μάνκα για τρία λεπτά. Κύριε Φεπουργέ, εκπρόσωπε τη Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι στο σχεδιασμό του προπολογισμού πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην βασική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον προπολογισμό. Οτιδήποτε δεν αφορά την νομοθετική μας αυτή, το νομοθετικό μας καθήκον για τον προπολογισμό θα πρέπει να μένει στο περιθώριο. Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή των Προπολογισμών και το Προεδρείο του Συγγελαγής του Κοινοβουλίου συναντήθηκαν και θέλω να ευχαριστήσω εδώ γιατί στην συνάντηση της Επιτροπής Προπολογισμού έγιναν δεκτές σημειώσεις που προτείναμε και η καλύτερη χρήση των δημοσιονομικών μας πόρων. Ωστόσο και πάλι υπάρχουν ελλείψεις και κενά. Δεν πετυχαίνουμε τα απαιτούμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά ιδίω τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ιδίω για την ασφάλεια και το κτίριο λόγου χάρη εδώ στο Στρασβούργο. Όπω ξέρετε, εδώ ερχόμαστε τέσσερι μέρε το μήνα και ω πρόσφατα τα κτίρια του Στρασβούργου φυλάσσονταν 365 ημέρες το χρόνο. Ε, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και η γραμματεία και το προσωπικό της το εντόπισαν αυτό και βρήκαμε τρόπο να γίνουν ε, οικονομίες, εξοικονόμηση τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επίσης, στον τομέα της μετάφρασης υπάρχουν κάποιες υπερβολές. Δεν υπάρχει κατάλληλη οργάνωση. Δεν υπάρχει η καλύτερη διάρθρωση των μεταφραστικών δυνατοτήτων. Τα θεσμικά όργανα που θέλουν μεταφράσεις πολλές φορές αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις μεταφράσεις αυτές χωρίς να κοιτάζουν αν υπάρχουν ε, διαθέσιμοι υπάλληλοι σε άλλα θεσμικά όργανα. Το 5% λοιπόν ε, του μεταφραστικού κονδυλίου θα μπορούσε να περνάει σε ένα αποθεματικό και να απελευθερώνεται όταν τα θεσμικά όργανα αποδεικνύουν ότι έχουν φτάσει στα όρια, των, ε, ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων τους. Θα εξοικονομήσουμε έτσι 11 εκατομμύρια ευρώ. Και επίση κατά του δημοσιονομικού ελέγχου. Συζητήσαμε χθε με τι πολιτικέ ομάδε και εκφράστηκε πολιτική βούληση να γίνει σωστή κατανομή των ελέγχων. Σε ό,τι αφορά το κονδύλι για τα κτίρια, αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Στο παρελθόν, τα, τα θεσμικό τα θεσμικά όργανα δεν ήταν πάντοτε αποτελεσματικά στην ενοικίαση, την αγορά και πώληση των κτηρίων. Σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, τα θεσμικά όργανα πάλι δεν συνεργάζονται μεταξύ του. Γι' αυτό ζητήσαμε από το διοικητικό προσωπικό να ασχοληθεί με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό τη αγορά και πώληση κτηρίων. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα χρειαζόμαστε ένα κοινό πρόγραμμα για την πολιτική των κτηρίων. Καλύτερη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Καλωσορίζω λοιπόν το γεγονό ότι το Συμβούλιο έχει εγκρίνει αυτό το στοιχείο ως μια προτεραιότητα. Ευχαριστούμε κύριε Μάνκα. Και τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, ο κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Σεμετά, μια που χθε επιβεβαιώθηκε ότι αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευχόμεθα να έχουμε την ίδια καλή συνεργασία όπως τον προκατοχό του και επίση του ευχόμαστε μια σταθεροδρομία πολιτική ε, το, το ίδιο επιτυχημένο όπως και Γκριμπασκάιτα. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια κρίση, από την προετοιμασία των ε, μεγάλων διπλωματικών ραντεβού και συναντήσεων και επίση πάρα πολύ μεγάλε σημαντικέ θεσμικέ αλλαγέ μέχρι και ακόμα και στου κόλπου τη Ένωση. Μέσα σε αυτή την περίοδο η Επιτροπή των Προπολογισμών θα προσπαθήσει να δείξει στάση να κρατήσει από πνεύμα συνεργασία και το είπε ο εισηγητή μα ε, καταδικάζουμε τι προτάσει του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με προτάσει τη Κομισιόν, Όμω καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση των δημοσιονομικών των κρατών μελών δεν επιτρέπει φέτο να προχωρήσουμε παραπάνω. Όσον αφορά την χρήση του 2010 για τον προπολογισμό, έχουμε ε, την υποχρέωση το να ε, ολοκληρώσουμε το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης με τη χρηματοδότησή του που ξεκίνησε και θα συνεχίσει το 2010. Όμως δεν θα πρέπει αυτό να είναι εις βάρος άλλων πολιτικών προτεραιοτήτων που ήδη έχουν κρυθεί και αποφασιστεί από κοινού, από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Πέραν όμως του 2010 θα ήθελε το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με Συμβούλιο και ε, Προεδρία με ε, Επιτροπή και με την επόμενη και με αυτή την Προεδρία όσον αφορά τους εξής άξονες. Πρώτα-πρώτα εάν τα πράγματα πάνε όπως ε, θέλουμε στην Ιρλανδία, να ξεκινήσει η διαδικασία του ενός χρονοδιαγράμματος, μιας μεθοδολογίας που, ε, θα αφορά την ε, θέση ισχύ της συνδίκης της Λισαβόνας. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση ε, ε, των, των πολιτών προγραμμάτων του Μαΐου του 2006 διότι σήμερα έχουμε την ε, οικονομική κρίση, έχουμε τις πάρα πολύ κρίσιμες εντάσεις στο ενεργειακό, στις πρώτες ύλες, αλλά και στα είδη διατροφής. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος επίσης. Δυστυχώς έχουμε και την ε, αυτή τη στιγμή αποτυχημένη στρατηγική της Λισαβόνας οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτόν τον πολιτή σχεδιασμό που τον χρειαζόμαστε και αυτό θα απασχολήσει την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση των ε, κοινοτικών πόρων Λόγω της κρίσης ε, τα κράτη-μέλη διστροπούν όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ευρώπης εμείς έχουμε πρόβλημα επομένως εδώ στην Ευρώπη, όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε κάτι για να υλοποιηθεί αυτή η, αυτό το σχέδιο της ανάκαμψης ε, και πώς θα φτάσουμε σε αυτή την χρηματοδότηση που θέλουμε εδώ και μια τετραετία ε, να μπορέσουμε να καθορίσουμε κάποιους άξονες εργασίας ώστε να ξεκινήσει αυτό το, το, το, το όραμα από του χρόνου ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαμασούρ, τον πρώτο τη Επιτροπή των Προπολογισμών, ο οποίο πάρα πολύ σαφώς μας ε, είπε την ε, θέση του Ευρωπαϊκού και τώρα θα δώσουμε τον λόγο στον ε, κύριο Υπουργό, τον κύριο Χάν Λίνμπλαντ, για να μας πει ε, τις θέσεις του Συμβουλίου. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε με προσοχή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας ανέφεραν ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τώρα το φθινόπωρο. Όμως έχουμε και άλλα, ίσως πιο δευτερεύοντα ζητήματα για φέτος το φθινόπωρο. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, πώς θα χρηματοδοτηθεί. δεν μπορούμε παρά να τρέφουμε ε, βάσιμες ελπίδες. Ε, πρέπει να πετύχουμε, καταδικασμένοι να πετύχουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, άλλη εναλλακτική. Γιατί υπάρχουν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, αλλά υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμοι. Και μακροπρόθεσμα εννοώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την πολιτική, για την αλλαγή του κλίματο. Εν πάση ευχαριστούμε. Δώσατε το λόγο. Ευχαριστούμε εμεί, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ όλου όσου έλαβαν το λόγο, λέει ο Πρόεδρο, και μην ε, δυσμονείτε ότι πρόκειται για μια αρχική ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τον προπολογισμό τη κρίση του 2010. Συγχαρητήρια επίση και στον ε, κύριο Επίτροπο για την ανάληψη των καθηκόντων του. Πρόκειται από την Λιθουανία και είμαι σίγουρο ότι η σταδιοδρομία σα θα είναι ε, πάρα πολύ καλή. Άλλωστε, έχετε ε, κρατήσει με επιτυχία το τιμόνι της πολιτικής της χώρα σας. Και τώρα πάμε παρακάτω στην ε, διάταξη που προβλέπει δηλώσεις του Συμβουλίου και της για τη μετανάστευση, το ρόλο της Frontex αλλά και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ο πρώτος αγορητής για σήμερα το πρωί θα είναι ο κύριος Τομπίας Μπίλτρομ ε, εκ μέρους του Συμβουλίου.